Συνεπώς έχει καθοριστεί η μερίσια διάταξη. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο σημείο δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκιόρη, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, αξιότιμα μέλη. Είναι η τελευταία φορά που μιλώ στην Ολομέλεια ενώπιον ε, στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας ε, και τον Ιανουάριο σας ε, υποσχεθήκαμε ότι θα έχουμε μία Προεδρία φιλική προς το Κοινοβούλιο. Γνωρίζοντας τις συνθήκες της συνθήκης της Λισαβόνας, Σα παρακαλώ, μπορείτε κάλλιστα να αποχωρήσετε από την αίθουσα, αλλά να μην ε, παρενοχλείτε του υπολείπου. Θα μπορούσατε ίσω να παραμείνετε και στην αίθουσα, δεδομένη και τη σημασία του θέματο που συζητάμε. Σα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε λοιπόν τι συνέπειε τη συνθήκη τη Λισαβόνα και γι' αυτό είχαμε και συνειδητοποιήσει ότι η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη τη θα ήταν υψής τη σημασία για την επιτυχία οποιασδήποτε προεδρία στο μέλλον. Οι Ευρωπαίοι πολίτες στρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αποτελέσματα, χωρί να ασχολούνται ιδιαίτερα με τη διάκριση μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου. Και έχουν δίκιο. Η ευθύνη μα είναι κοινή και το ίδιο έχουμε κοινή ευθύνη για την επιτυχία και την αποτυχία. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Γι' αυτό λοιπόν η συγκεκριμένη συζήτηση αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία να δούμε τι επιτεύχθη για πολλά θέματα σε στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχά, να ξεκινήσω με την οικονομική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έτσι, σε ένα κύκλο πολιτικής έχουμε τους δύο βραχίονες της οικονομικής ανάκαμψης. Την χρηματοπιστωτική σταθερότητα που, που βασίζεται στην δημοσιονομική σταθερότητα και αντικατοπτρίζεται στη σταθερότητα και σε προγράμματα σύγκλησης και διαθροτικών μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις πιο ευάλωτες ομάδες. Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και κρατών μελών για την ε, εφαρμογή ε, των προγραμμάτων μεταρρύθμισης και των συστάσεων, το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο διέκρισε ένα εξάμεινο μόνο και ούτε στιγμή παραπάνω. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προσκληθεί να ε, εγκρίνει τι συγκεκριμένε συστάσει αναχώρα που ενεκρίθησαν από το Συμβούλιο και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ε, τι ε, αποφάσει που ελήφθησαν από όλα τα κράτη-μέλη για τον προπολογισμό και τι διορθωτικέ μεταρρυθμίσει του. Να σας πω επίσης ότι και στις τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουμε μία αναφορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ώστε να μπορεί να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Όσον αφορά το σύμφωνο Ευρώ-ΣΥΝ, πολλά από τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν παρουσίασαν δεσμεύσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου 100 διαφορετικά μέτρα. Αυτές οι δεσμεύσεις αποτελούν ένα καλό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του συμφώνου που πλέον πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, ο βαθμός της φιλοδεξίας και ακρίβειας αυτών των αρχικών δεσμεύσεων είναι άνισος. Κατά την προετοιμασία των επόμενων δεσμεύσεων, τα κράτη-μέλη θα διασφαλίσουν ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογή, μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση και έναν υψηλότερο βαθμό φιλοδοξία. Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στι έξι νομοθετικέ προτάσει για την οικονομική διακυβέρνηση, το πακέτο των έξι όπω το αποκαλούμε. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, διότι βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη τη Ολομέλεια. Θα ήθελα απλώ να σα υπενθυμίσω ότι η Ουγγρική Προεδρία είχε λάβει την εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Μετά από την υιοθέτηση μιας γενικής προσέγγισης από το Συμβούλιο το Μάρτιο, αρχίσαμε αμέσω τις εργασίες και ε, ξεκινήσαμε εντατικέ ε, τριμερεί διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τρία θεσμικά όργανα έκαναν εξαιρετικό έργο. Η αρχική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε περίπου 2.000 τροπολογίες. Πλέον έχουμε καταφέρει να, μειώ, ε, να μειώσουμε τις εκκρεμότητες σε ένα μεγάλο σημαντικό θέμα και κάποια τεχνικής, ε, τεχνικά ζητήματα ίσονος σημασίας. Είμαι προσωπικά πεπισμένη ότι το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πιο στεναρό και είναι καταλληλότερο για την πρόληψη ε, μελλοντικών κρίσεων. Θα ενημερώσουμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναλόγως και έτσι θα αναφέρουμε στο όργανο το οποίο μας ανέθεσε αυτή την αποστολή. Εγώ προσωπικά ε, έκανα συναρπαστικές συζητήσεις με πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου και δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την εμπειρία. Επειδή είμαστε μια Προεδρία φιλική προς το Κοινοβούλιο, ελπίζουμε τα αποτελέσματα τα οποία μας οδήγησαν στη, στα πρόθυρα της συμφωνίας να μην ε, έγιναν επιματέω. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυρίως οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν να επιδείξουμε ευθύνη, αποφασιστικότητα και να δράσουμε ε, κατά των χρεών που είναι το βασικό πρόβλημα των οικονομιών μας. Τέλος, σημειώνουμε επίσης ότι το θέμα της Ελλάδος θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα τώρα να περάσω στα θέματα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με το άσυλο, τη μετανάστευση και τη Σέγγεν βάσει των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων στι 9 Ιουνίου του 2011. Εν ώψη και των ε, πρόσφατων εξελίξεων, το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο θα συζητήσει ιδέες και θα δώσει περισσότερη πολιτική καθοδήγηση και συνεργασία στον τομέα Σέγγεν. Θα συζητήσει και κάποια θέματα ε, σχετικά με ένα πιθανό μηχανισμό διασφάλισης. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι η καλή λειτουργία του Σέγγεν απαιτεί να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη πλήρως τους κανόνες και έτσι να ενισχυθεί και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ε, ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Να αναφερθώ τώρα στην ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων. Πρόκειται για ένα διαφορετικό κεφάλαιο του κοινοτικού κεκτουμένου ε, σε σχέση με τη Σέγγεν, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Και τα δύο είναι από τα πιο προφανή και πιο δημοφιλή επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν και έχουν κάθε πρόθεση να τα διαφυλάξουν. Η λογική που διέπει τη Σέγγεν δεν έχει αλλάξει. Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική διαχείριση για να μπορούμε όλοι να ταξιδεύουμε χωρίς ελέγχους ε, στην περιοχή Σέγγεν. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις για το κανονισμό τροποποίησης της Frontex. Η Frontex είναι το βασικό εργανείο στα χέρια μας, ε, ικανή και αναγκαία συνθήκη για να ελέγχουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Η Προεδρία χαιρετίζει τα πολύ θετικά αποτελέσματα των προσφάτων συνομιλιών. Τα κράτη-μέλη συζητούν σήμερα το απόγευμα τα αποτελέσματα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία εν ευθέτω χρόνο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, οι πρόσφατες εξελίξεις ε, ε, έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Χρειαζόμαστε ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη προστασίας. Πρέπει λοιπόν ε, το κοινό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2012 βάσει προτύπων υψηλής προστασίας καθώς και δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών που θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις καταχρήσεις και θα επιτρέψουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων ασύλου για να μπορέσουμε να έχουμε βιωσιμότητα του συστήματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δει επίσης και τι δυνατότητες υπάρχουν για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ο στόχος είναι να βρούμε να, τη ρίζα του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να αναπτύξουμε εταιρικέ σχέσεις με τις χώρες της νότιας γειτονίας. Ως πρώτο βήμα θα υπάρξει ένας ευρύτερος διαφρομένος διάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια με στόχο να έχουμε απτά ωφέλη για αυτά αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, κάποια πράγματα για την Κροατία. Ε, μετά από τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία, που θεωρήθηκε μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας, ε, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, στην οποία θα πρέπει να ο φόρο τιμής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις ε, προσχώρησης με την Κροατία μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2011 και η υπογραφή της ε, συνθήκης προσχώρησης προβλέπεται πριν από το τέλος του έτους. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια νέα όθηση για την ευρωπαϊκή προακτική των Δυτικών Βαλκανίων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξανασυζητήσει το ζήτημα αυτό το Δεκέμβριο του 2011 και θα χαιρετήσει κατά πάσα πιθανότητα και τη σύλληψη και τη μεταφορά του στρατηγού Μλάντιτ η Σερβία έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προς την ευρωπαϊκή προσχώρηση. Για την νότια γειτονία Θέλουμε να ε, υιοθετήσουμε μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις με τις γείτονες χώρες, η οποία συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρες, ε, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις ε, σε κάποια τμήματα της, ε, των χωρών της Νότιας Γειτονίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει και μια δήλωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και για την διορισμό του Μάριο Ντράγκη ως ε, τον επόμενο διοικητή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τέλο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα θα εγκρίνει και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη και θα ανασχοληθεί με το θέμα των Ρωμά και έτσι υλοποιούνται δύο περαιτέρω προτεραιότητε τη Ουγγρική Προεδρία. Η στρατηγική για το Δούναβη θέλει να ενισχύσει τι δυνατότητε μια ολόκληρη περιοχή να εναγκαλίσει τη διαφοροποίηση των κρατών μελών με τρίτε χώρε ε, στα δυτικά Δαλφα... Ε, Δαλκάνια, ε, λαού και κοινότητε στα πλαίσια των στρατηγικών για τους Ρωμά θα έχουμε για πρώτη φορά ε, μια εξαιρετική ευκαιρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι είχατε μια εξαιρετική έκθεση που ε, αποτέλεσε και πάρα πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας στο Συμβούλιο. Η Ευρώπη θα αποδείξει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Ορμπάν, έχει και καρδιά και όχι μόνο μυαλό. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη, η Ουγγρική Προεδρία επέλεξε την ισχυρή Ευρώπη ως σύνθημά της. Α εκφράσω την ελπίδα ότι θα συμφωνήσετε και εσείς με την άποψη του Προέδρου Μπούζεκ, ο οποίος είπε πρόσφατα ότι μετά την Ουγγρική Προεδρία η Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ εκ βάθους καρδίας για τη συνεργασία σας ε, στο περασμένο εξάμεινο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον Πρόεδρο Μπαρόζο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Το Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει πάρα πολύ ουσιαστική ημερήσια διάταξη η κυρία Υπουργό, εδώ πέρα εκπροσωπεί το Συμβούλιο και θέλω να την ευχαριστήσω για την δέσμευση την οποία απέδειξε αυτού του έξι μήνε και θα ήθελα να εστιαστώ σε ορισμένα ζητήματα. Απέθυνα μία επιστολή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζοντα τι θέσει τη Κομισιόν στα σημαντικότερα θέματα τη ημερήσια αυτής διάταξη και θέλω να μοιραστώ αυτέ τι θέσει μαζί σα τέλο θα κάνω και κάποια σχόλια για την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο θα κάνει σημαντικά βήματα για να διασφαλίσει πως η λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής είναι και σαφέστερη και αποτελεσματικότερη. Πρώτα απ' όλα έχουμε το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά το Κοινοβούλιο για την εξαιρετικά σκληρή δουλειά και δέσμευση που έχει επιδείξει στην διατήρηση υψηλού επίπεδου φιλοδοξίας για το ζήτημα αυτό. Αργότερα, σήμερα το απόγευμα, ο Επίτροπος ο κύριος Ρεν θα εκφράσει την ε, λεπτομερή μας θέση για το εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα. Να σας πω τώρα πως αναμένω να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη με το Κοινοβούλιο, γιατί η οθέτηση του πακέτου αυτού είναι σημαντική για την ολοκληρωμένη απάντησή μας στην κρίση. Συμφωνία από το πακέτο αυτού είναι ζωτική και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες πως τη στιγμή που προσπαθούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις τέτοιου μεγέθους δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε στους θεμελιώδεις πυλώνες απάντησης σε αυτή την κρίση. Θεωρώ πως η συμφωνία σε αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τους μηχανισμούς οικονομικής υποπτίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ικανότερη να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις δημοσίων χρέων και ελλημάτων που δεν μπορούν να είναι βιώσιμα καθώς και των βλαβερών δημοσιονομικών ανισορροπιών. Και βέβαια η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Θα έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε επίση τυχόν καταστάσει που θα προκύψουν. Δεύτερον, αναμένω από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων να υιοθετήσουν τις συστάσεις αναχώρα που παρουσίασε η Κομισιόν στις 7 Ιουνίου. Είναι, όπως ξέρετε, η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συστάσεις βασίζονται σε εκτεταμένη ανάλυση από την Κομισιόν των σχεδίων των κρατών μελών για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση ταυτόχρονα με υγιή δημόσια οικονομικά. Είναι στέλιε εστιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα. Βεβαίω οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη ήταν πάρα πολύ έντονε μερικές φορές, αλλά είμαι ικανοποιημένος για το ότι το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει αρκετά φιλόδοξο. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αφενός να εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς και από την άλλη να αγνοούμε μια άφρονα οικονομική πολιτική. Οπότε αναμένουμε βεβαίως και συγκεκριμένες συστάσεις που θα έρθουν από την Κομισιόν αναχώρα. Πρόκειται επίσης ε, για μια προσέγγιση η οποία προτείνει περισσότερη οικονομική ευθύνη γιατί βεβαίως ο οικονομικός αυτός χώρος είναι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των οικονομιών μας. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την αλλαγή της συνθήκης η οποία είναι απαραίτητη για τον ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα από το 2003 με τη δυνατότητα που θα έχει να στηρίζει τα κράτη-μέλη σε οικονομικές δυσκολίες με βάση αυστηρού όρους. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερότητα μαζί βεβαίω με την αυξημένη δανειοδοτική ικανότητα του μηχανισμού ε, δημοσιονομικής ε, σταθερότητας θα έχουν στόχο να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά. Θα θυμάστε επίσης πως τον Ιανουάριο στην έκθεσή μας περί ανάπτυξης είχαμε τονίσει την ανάγκη το EFSF να έχει την δυνατότητα να δανείζεται. Μας είχαν ασκήσει τότε μεγάλη κριτική, αλλά τώρα ομόφωνα οι κυβερνήσεις της Ευρώπης αποφάσισαν να αυξήσουν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα δανεισμού. Μα ρωτιέμαι μήπως θα ήταν δυνατό να έχει εγκριθεί πριν από μερικούς μήνες ήδη το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης, οι συστάσεις αναχώρα και ο μηχανισμός σταθερότητας, αυτή είναι ακριβώς η αντίδραση της Ευρώπης και θα πρέπει να βγάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα από αυτή την κρίση και να δράσουμε αναλόγως. Για να απαντήσουμε στην οικονομική κρίση πρέπει να συνεισφέρει ο κάθε κλάδος και πολύ περισσότερο ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Υποσχέθηκα στο Κοινοβούλιο πως η Κομισιόν θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για έναν φόρο στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Θα έχει τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να αποφυχθεί ο κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μη συντονισμένα εθνικά φορολογικά μέτρα. Δεύτερον, ο φόρος αυτός έχει στόχο να δημιουργήσει αντικίνητρα για υπερβολικά επικίνδυνες ή καθαρά κερδοσκοπικές συναλλαγές. Τρίτον, να διασφαλίσουμε πως ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνεισφέρουν με τρόπο δίκαιο και ουσιαστικό στην αντιμετώπιση της κρίσης καθώς και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες για τα υπερβολικά κέρδη. Τα πολύ υψηλά μπόνους που εξακολουθούν να πληρώνουν οι τράπεζε στου τραπεζίτες, τους οποίους διασώσαμε με τεράστια ποσά δημοσίου χρήματο, υποδεικνύουν πω υπάρχουν υπερβολικά κέρδη στον τραπεζικό τομέα και πω και αυτό ο τομέας θα πρέπει να συνεισφέρει στο κοινό καλό. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η μετανάστευση. Το ζήτημα αυτό ήρθε στο προσκήνιο του τελευταίου μήνε, ειδικά υπό την πίεση των ε, γεγονότων στην Νότια Μεσόγειο. Μίλησα το Μάιο στο Κοινοβούλιο για το μεταναστευτικό πακέτο της Κομισιόν, το οποίο βάζει όλες τις πρωτοβουλίες αυτές σε ένα πλαίσιο που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη να διαχειριστούν τη μετανάστευση και την κινητικότητα επικών τρίτων χωρών σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η μετανάστευση, ας το αντιμετωπίσουμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ανακοινεί τα πάθη, αλλά η Κομισιόν δεν θα ανοιχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια να υπονομευθούν οι αρχέ τη Σέγγεν. Μάλιστα, επιζητούμε ακριβώ το αντίθετο μέσω μια ενίσχυσης Ευρωπαϊκή προσέγγιση και τη ελεύθερη διακίνηση. Η Κομισιόν πρότεινε να ενισχυθεί η διακυβέρνηση τη ε, περιοχή Σέγγεν και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των κρατών μελών στη διαχείριση των εξωτερικών μα συνόρων. Αυτό θα γίνει και μέσω της ενίσχυσης της Frontex και μέσω ενός μηχανισμού αξιολόγησης όπου θα συνεργάζονται οι Εθνικές Υπηρεσίες Συνοριοφύλαξης. Επίσης, κοιτάμε ένα σύστημα ρητρών διασφάλισης που θα επιτρέπει την υιοθέτηση αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν πιθανές δυσκολίες όπου τα κοινά εξωτερικά μας σύνορα υφίστανται τρομερές πιέσεις ή όπου τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις ελέγχου των συνόρων τους. Οι αποφάσεις για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης κάθε κατάσταση θα λαμβάνονται σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην υπάρχουν μονομερείς ενέργειες των κρατών μελών και θα μπορούσε να προβλεφθεί ως τελευταία λύση και αν το δικαιολογεί η κρίσιμη κατάσταση την προσωρινή επανεισαγωγή εσωτερικών ε, ελέγχων στα σύνορα πάντα στο κοινοτικό πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει πως πάει προς τα πίσω η εξέλιξη των συνόρων, ενισχύουμε την ευρωπαϊκή διάσταση του συστήματος έτσι ώστε να μην αισθάνονται τα κράτη-μέλη πίεση να δράσουν μονομερός. Θα αναμένω στήριξη αυτών των προτάσεων από το Συμβούλιο για να οριστικοποιηθούν και να έχουν ευκαιρία να επιτύχουν. Το πακέτο της μετανάστευσης θα ολοκληρωθεί με προτάσεις για κοινό αποτελεσματικό σύστημα ασύλου που θα εγγυάται σε όσους ζητούν άσυλο ή συμμεταχείριση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι σίγουρος πως Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα υιοθετήσουν τις προτάσεις Κομισιόν για ελάχιστες προδιαγραφέ για υποδοχή ετούντων άσυλο και ετούντων καθιστώτο πρόσφυγα. Ζητάω, θα ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εθετήσει αυτό το πακέτο το συντομότερο δυνατόν εντός ε, της συμφωνηθής προθεσμίας. Επίσης το Συμβούλιο θα, ζητήσει, θα συζητήσει την Ευρωπαϊκή Γειτονία, ειδικά τα ζητήματα δημοκρατίας και της ε, κοινή ευημερία με την Νότιο Μεσόγειο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εταίρους μα που κοιτούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη της δημοκρατικής μετάβασης αυτής και δεν πρέπει να του απογοητεύσουμε. Ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η σύσταση της Κομισιόν έτσι ώστε η Κροατία να γίνει το 28ο κράτος μέλος μέχρι ελπίζουμε την 1η Ιουλίου 2013. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να υπογράψουμε την λήξη των υπολείπων κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις. Δύο λόγια για την Ελλάδα, γιατί βεβαίω ελπίζω και τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν στο υψηλότερο επίπεδο την κατάσταση αυτή, που βεβαίω είναι σοβαρή όχι μόνο για ένα κράτο μέλο, αλλά για τη σταθερότητα τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα τη Ελλάδα θέτει πολύ σημαντικά θέματα, όχι μόνο όσον αφορά την νομισματική σταθερότητα, αλλά όσον αφορά και τι κοινωνικέ δεσμεύσει και την πολιτική αποφασιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων επιτρέπει στην ε, κυβέρνηση να δημιουργήσει συνένεση στήριξης του μεταρρυθμιστικού πακέτου που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ για φορολογικά μέτρα, ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην ανάπτυξη. Γιατί ας είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο σχέδιο αυτό, οπότε ας ξεκινήσουμε να δρούμε. Ξέρω πως πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα περνάνε μεγάλες δυσκολίες και έχουν αβεβαιότητα. Το μήνυμά μου στον ελληνικό λαό είναι πως εάν η κυβέρνηση δράσει η Ευρώπη θα βοηθήσει. Εάν η Ελλάδα μπορεί να δείξει πως πραγματικά είναι δεσμευμένη στο μεταρρυθμιστικό πακέτο που έχει συμφωνήσει με Ευρωπαϊκή Ένωση και του, θα συνοδεύσουμε την Ελλάδα στην πορεία τη στην ανάπτυξη. Γιατί η η εξυγίανση των νομικών είναι απαραίτητη, αλλά ο στόχος είναι η ανάπτυξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα ευρώ που ξοδεύεται σε τοκοχρεολύσια δεν πηγαίνει, το στερείται ο ελληνικός λαός. Οπότε θα πρέπει να μειωθεί το χρέος και να ελεγχθεί το έλλειμμα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία για να υπάρξει ανάπτυξη. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός πως αντιμετωπίζοντας τόσο δύσκολες συνθήκες είναι αναγκαία εθνική συνένεση. Εθνική συνένεση και όχι μικροκομματική πολιτική. Χρειάζεται εθνική συνένεση στην Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών η Ελλάδα για τις πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Δευτέρα βράδυ συναντήθηκαμε με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου και συζητήσαμε μια πιο στρατηγική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υψηλά ποσά υπό την πολιτική συνοχή και θεωρώ πως θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης και να επιταχυνθεί η απορρόφηση αυτών των ποσών για να βελτιωθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα. Αυτό θα γίνει με τα υπάρχοντα ταμεία, θα είναι ένα συνολικό πρόγραμμα τεχνικής αρροχής, που θα εστιάζεται στην ανάπτυξη και στις δουλειές, αλλά με χαρακτήρα κατεπηγόντος. Γιατί όπως σας είπα η Ελλάδα βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση. Θα συζητήσω με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα. Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση μπορεί να καταβάλει αυτές τις προσπάθειες. Αλλά θα πρέπει όσοι μπορούν να βοηθήσουν να το κάνουν. Δηλαδή τεχνική αερογή από όλα τα κράτη-μέλη. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση και θα πρέπει να είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει και να συνεχίσει αυτή τη θετική πορεία πάντα με τους αυστηρούς όρους που έχουμε θέσει για τη μεταρρύθμιση. Το σχέδιο το μεταρρυθμιστικό απαιτεί εξαιρετικές προσπάθειες από τον ελληνικό λαό και η Κομισιόν προτείνει μια εξαιρετική απάντηση για να δείξουμε στον ελληνικό λαό πως κάνουν θυσίες, γνωρίζουμε πως κάνουν θυσίες, αλλά στο τέλος αυτής της πορείας υπάρχει ελπίδα και οι λύσεις είναι πραγματικά εφικτές. Κάνουν περικοπές σημαντικές, αλλά είναι απαραίτητες αυτές για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι η απάντηση και θα συνεργαστούμε με τις ελληνικές αρχές και τον ελληνικό λαό για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Μπαρόζο. Να δώσω τώρα το λόγο στους αγορητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντόλ, ο οποίος έχει πέντε λεπτά στη διάθεση. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί Ενικό πρώτα απευθύνω σε εσάς, σε σένα, δύο λόγια ευχαριστίες για όλη τη δουλειά και τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκες με τη δουλειά αυτή και κυρίως συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Οφείλουμε νομίζω να το πούμε. Ε, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά θερμά. Μα τη χειροκροτάτε φυσικά, δεν θα μπορούσαμε τίποτε άλλο να κάνουμε αφού ξέρουμε ότι μέσα από τη δική μας την πολιτική ομάδα ξεπετάχτηκε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν προκύπτει μέσα σε πλαίσιο και σε δεδομένα από μεγάλη ένταση. Με ένταση και σε επίπεδο κοινή γνώμη μεταξύ των κρατών μελών, ε, ε, τη κοινή γνώμη στα κράτη-μέλη, σε σχέση με τι καυτέ απαντήσει ε, και την ανταπόκριση σε αυτέ, τη διακυβέρνηση λοιπόν την οικονομική και τη μεγάλη κρίση, τώρα την κρίση του ευρώ. Στην Ελλάδα ιδιαίτερω, αλλά και σε όλα τα κράτη, αισθάνεται βαθύτατο άγχο, ανησυχία, φόβο για το μέλλον του πολίτη, όπω και για το μέλλον των παιδιών του. Και επί ευκαιρία ήθελα να απευθύνω τρία μηνύματα προς τους Έλληνες φίλους. Πρώτο μήνυμα, η Ευρώπη είναι αλληλέγγυα προς την Ελλάδα και κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς οι Ευρωπαίοι για να σας βοηθήσουμε να βγείτε από μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη με συνθήκες ευθύνης και αλληλεγγύης και επιμένω στη λέξη ευθύνη. Δεύτερο μήνυμα, η κατάσταση που διαβιώνουν οι Έλληνες, που βιώνουν οι Έλληνες είναι αποτέλεσμα μεγάλου χρονικού διαστήματος στο οποίο ζούσαν με δαπάνε υψηλότερε από αυτέ που επέτρεπαν τα μέσα του, όπω άλλωστε πολλά άλλα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να το πούμε και καλό του Ευρωπαίου να δουν την αλήθεια κατάματα. Το τρίτο μου μήνυμα αποτελεί απόρρια των δύο πρώτων. Η Ευρώπη δεν μπορεί να στηρίξει, να βοηθήσει την Ελλάδα, όπω και κάθε άλλο κράτο που αντιμετωπίζει δυσκολία, παρά μόνο αν αυτή αναπτύξει κάθε δυνατό μέσο και μέσο στη διάθεσή τη, έτσι ώστε να εξηγειάνει την οικονομία τη. Αυτό περνάει και μέσα από τι θυσίε, αλλά ταυτόχρονα και μακροπρόθεσμα θα προσφέρει θετικέ εξελίξει για τη χώρα. Και έτσι πρέπει να πω και θα πρέπει να αναφερθώ στο παράδειγμα της Λετωνίας, η οποία έχει φτάσει στα πρόθυρα της πτώχης πριν από μερικά χρόνια και χάρη στον Πρωθυπουργό Ντομπρόφσκι και το ε, πρόγραμμα εξυγίανσης ε, που ακολούθησε αυτός μπόρεσε να διασωθεί. Δύο στάσεις διαφορετικές και εναλλακτικές πιθανέ πιθανές ε, μπορεί να αναπτύξει κανείς έναντι της κρίσης. Μπορεί κανείς να κατεβαίνει στον δρόμο, να κάνει απεργία, δικαίωμα συνδικαλιστικών και εγώ συνδικαλιστή που είμαι στο παρελθόν, είτε εκφράζοντα με την ανησυχία του να ανασκουμποθεί και να κάτσει να δουλέψει για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση με σωστέ πολιτικέ. Η ομάδα μου, κυρίε και κύριοι, απευθύνει έτοιμα για υπέρβαση, για ανάληψη συνείδηση στι χώρε μα ότι τα μέτρα αυτά είναι σκληρά, μεν αλλά απαραίτητα. Με το να ανακηρύσουμε από τον Πομπέου Στράγο στην Ευρώπη το Διεθνέ Πραγματικό Ταμείο κάποιων άλλων, δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. και εμείς σημαίνει και η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη αλλά και κάθε Ευρωπαίος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βγούμε από την κρίση με μεγάλες και βαθιές μεταρρυθμίσεις της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό αναμένουμε. Το ευρώ είναι το μεγάλο νόμισμα, το ενιαίο νόμισμα και η έκφραση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, αλλά το τμήμα της οικονομικής ενοποίησης είναι να επαρκέσει και σε αυτό πληρώνουμε το βαρύ τίμημα. Έτσι λοιπόν η ομάδα μας καλεί, απευθύνει έκκληση για μια μεγάλη μεταρρύθμιση οικονομική έτσι ώστε να μπορούμε να μην, να μην επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να διαφεύγουν των υποχρεώσεών τους, να απαλλάσσονται εύκολα από τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε με την πρώτη ευκαιρία παρεκκλήσεις από, τα, από τους κανόνες που επιβάλλουμε. Αυτό είναι και ένα από τα διδάγματα που μας έχει φέρει η κρίση. Να διδαχθούμε από τα σφάλματα του παρελθόντος μπορούμε, μπορεί να μας οδηγήσει προς καλύτερο μέλλον. Και έτσι προχωρώντα το θέμα τη μελλοντική προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να είναι σε μερικού μήνε το 28ο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτή αποτελεί το επιστέγασμα των μεγάλων προσπαθειών του λαού τη Κροατία και τη κυβέρνηση του, που θα ήθελα να χαιρετήσω για τι προσπάθειε που κάνουν προ το κοινό καλό. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μεγάλε προσπάθειε και με ανταμοιβή αυτών οι αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός του άλλου, της ανθρώπινης αξίας, του πιο αδύναμου, της μειονότητας, πρέπει πάντοτε να προασπίζονται μέσα στην, στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, εκεί όπου το κέρδος μερικές φορές φαίνεται να επικρατεί σαν αρχή. Εάν ξεφύγουμε από το λαϊκισμό, εάν ξεφύγουμε από το εύκολο κέρδο, μπορούμε πιστεύω να προχωρήσουμε προ ένα καλύτερο μέλλον και ελπίζω αυτό το μέλημα να καθοδηγήσει του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων πάνω από οποιοδήποτε άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόλ και τώρα το λόγο στον κύριο Μάρτιν Σούλτ για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι. Σπάνια σπάνιστερη ήταν οι περιπτώσει όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε να συζητήσει προετοιμασία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνθήκε χειρότερε από αυτέ τη τωρινή κρίση και νομίζω ότι δεν έχει κανεί ψευδεστήσει πλέον. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό έχει ιστορική σημασία. Ιστορική σημασία γιατί λαμβάνει αποφάσει και για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εβδομάδα διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ε, χωρίο σε μια, ευρωπαϊκή, σε μια γερμανική ε, εφημερίδα όπου έλεγε στο άρθρο ότι ο Ευρωπαίος πολίτης δυσπιστεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τη έχει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Ο πολίτης στην Ευρώπη δυσπιστεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματά του. Είμαστε μέσα σε μια βαθιά κρίση, σε μια κρίση πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι γνωστά τα προβλήματα, Έχουμε όλοι αυτή την κόπωση από την κρίση. Από την κρίση. Το θέμα είναι αν μπορούμε να δώσουμε τα ε, σκληρά, σκληρές απαντήσεις που χρειάζονται. Αν έχουμε το θάρρος και την παρησία να τις ε, προβάλλουμε αυτές τις απαντήσεις ή αν από, από αδράνεια θα, θα αφήσουμε τις εξελίξεις να μας ξεπεράσουν. Και θα ήθελα να πω γιατί το πιστεύω βαθύτατα, ότι αυτό θα μας βάλει από την κρίση, ότι από αυτές τις συνθήκες δεν χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη, περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε το θάρρος και την παρησία, την κρίση, την παρούσα, να την διαχειριστούμε χάρη σε περισσότερη Ευρώπη. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Το συμβόλαιο αυτό, η Σύνοδος Κορυφής, θα ασχοληθεί, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα πρέπει να ανακτήσουν την δυνατότητα να διαχειριστούν τα, τα κράτη τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν αποφασίζουν πλέον αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το τι συμβαίνει μέσα σε ένα κράτος, αλλά οι 43 μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν μερικές φορές πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ ε, μάλλον ε, κεφάλαιο η αξία οικονομική από το ΑΕΠ της Πολωνίας. Άρα είναι ισχυρότεροι οι ε, διοικητές αυτών των ε, επιχειρήσεων, των 43 επιχειρήσεων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, Φερρυπίν. Και... Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι μηχανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προβαίνουν την παραμονή ακόμη ενός Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ σε κρίση και υποβάθμιση κατά μία, δύο, τρεις μονάδες κρατών της ζώνης του ευρώ. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοποιητικής ε, δυνατότητας, ποιοι είναι αυτοί, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι, κάποια συμφέροντα εκπροσωπούν και για κάποιες προτάσεις αξιολόγησης παίρνουν και τη σχετική αμοιβή, το αντίτιμο. Πρέπει λοιπόν να ανακτήσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το δικαίωμα στη δημοκρατική δράση, στη δημοκρατική διακυβέρνηση. Αυτό μπορούν να το καταφέρουν μόνο αν είναι ενωμένοι. Δεν μπορούν να το καταφέρουν αν ο καθένα κοιτάει σε διαφορετική κατεύθυνση. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού στα 27 κράτη-μέλη της. και έχουμε προβλέψεις δημογραφικές ότι μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια θα έχουμε μόνο 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν θα μπορούμε λοιπόν μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, τις νέες δυνάμεις που αναδύονται, τις ε, νέες οικονομίες που ενισχύονται. Δεν είναι δυνατόν από τη Μεγάλη Γερμανία μέχρι τη πιο μικρή Πάλτα να περιμένουμε, να κατακαιρματιστούμε και να διαλυθούμε. Θα πρέπει μόνο σε μια μεγάλη ένωση και δια, διυπηρωτική αντιπαράθεση να υψώσουμε το ανάστημα, ανάστημα τόσο στο θέμα του περιβάλλοντος όσο και στο θέμα της οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης μόνο εάν είμαστε ενωμένοι και αν έχουμε το θάρρος να σταθούμε ως η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου γιατί αυτό είναι η Ευρώπη και μπορεί να στεφθεί με επιτυχία αυτό το μεγάλο εγχείρημα μόνο εάν είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας. γιατί ισχύς εν και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα όχι απλώς φόρος χρηματοπιστωτικός φόρος αλλά φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όταν πουλάω γάλα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να πληρώσω φόρο προσθέμενης αξίας. Όταν, όταν πουλάω χρηματοπιστωτικό προϊόν πρέπει και εκεί πάνω να πληρώνω κάποιο φόρο. Δηλαδή φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι τα δεδομένα όλα επιτάπητος τα βλέπουμε ξεκάθαρα. Και ή θα τα καταφέρουμε με την ενότητα στην Ευρώπη και όχι με το να παίζει παιχνίδια εις βάρος του ενός κράτου το, κράτους στο άλλο και όχι με το να υπάρχουν αντιπαραθέσεις και εντάσεις μεταξύ μας. Μόνο ενωμένοι λοιπόν και για αυτό το λέω διότι η Ευρώπη είναι σε κίνδυνο και πολύ συγκεκριμένο κίνδυνο. Διότι εάν αποτύχει ως υπερεθνικό εγχείρημα η Ευρώπη, εάν καταρρεύσει η Ευρώπη κυρίες και κύριοι, δεν, δεν καταραίει μόνο μια πολιτική ενότητα. Ξυπνάνε πάλι τα παλαιά δαιμόνια, τα δαιμόνια του 20ου αιώνα, εκείνα που μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Η διάλυση της Ευρώπης σημαίνει διάλυση και εξαφάνιση μιας πολύ μεγάλης ιδέας. Ευχαριστώ. Πριν